θεωρηθεί ότι εγκρίνεται για ένα διορθωτικό που στην Ολομέλεια κατά την 24η ε, Ιουνίου σύμφωνα με το άρθρο 231 του κανονισμού γνωστοποιήθηκε δεν υπευλήθη έτοιμα για ε, ψήφιση και έτσι θεωρείται ότι το διορθωτικό αυτό εγκρίθηκε. Μπορείτε